216 αν εντό 24 ωρών δεν θέσει κάποια ομάδα ή τουλάχιστον 40 βουλευτές κάποια αντίρρηση θα τεθούν ε, θα εγκριθούν οι προτάσεις της Επιτροπής ε, Νομικών Θεμάτων. Επίση, ε, σύμφωνα με το άρθρο 74, συνυπέγραψαν τον Πρόεδρο του Συμβουλίου δύο νομικές πράξεις Σύμφωνα με την τακτική νομοθετική διαδικασία, οι τίτλοι θα δημοσιευθούν στα πρακτικά αυτής συνεδρίασης.